to start. We have just one hour, less than one hour actually. Ο Πρόεδρος. Βολτιέρη, έχουμε τώρα πάρα πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Είναι κάτι που το περιμέναμε πολύ καιρό και τελικά μπορέσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Επομένως θα πρέπει να ευχηθούμε το καλωσόρισμα στον ε, αντιπρόεδρο Μοσκοβησία αλλά και στον επίτροπο Ντομπρόφσκης και ε, τη σήμερα ημέρα, το, Μάρτιο του 18 θα πρέπει να συζητήσουμε και τη δεσμή των μέτρων τη 6η Δεκεμβρίου όσον αφορά την εμβάθυνση τη Νομισματική Ένωση. Αλλά επίση έχουμε και τι ε, εν εξελίξει σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει Οπότε περιμένουμε ανυπόμονα λοιπόν να σας ε, ακούσουμε και τον Μάιο έχουμε την επόμενη δόση αυτών των ε, μέτρων. Οπότε θα έχουμε και το Συμβούλιο του Ιωνίου, οπότε ελπίζουμε ότι θα έχουμε απλώ μια μετάθεση της προβληματικής για το επόμενο Συμβούλιο. Οπότε, πολλές, οπότε ε, φαίνεται μάλλον ότι πάει προς τα εκεί το πράγμα χωρίς να αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και Έχουμε όλες αυτές τις σημαντικές προτάσεις για τον ESM τη στατική σας για συντονισμό και διακυβέρνηση να μας πείτε πώς βλέπετε τις μελλοντικές εξελίξεις, πώς βλέπετε τις σκοπούμενες αλλαγές στον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις Ε, που θα έχει πιλωτικό χαρακτήρα. ούτως ώστε να έχουμε αναβάθμιση της προσπάθειας για τις επιθυμητές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους μακροοικονομική δυνατότητα σταθεροποίησης, εξυγίανση των δημοσιονομικών, Γι' αυτό και έχουν ε, κομικό χαρακτήρα οι προτάσεις σας. Ε, και τώρα πια φτάσαμε Μάρτιο ε, να συζητήσουμε αυτά τα μέτρα που προτάθηκαν τον Δεκέμβριο. Για να δούμε τι εξελίξει θα έχουμε τώρα Ζώνα αφορά αυτή τη δέσμη μέτρων. Πολιτικές μόνο παρατηρήσεις μπορούμε να διατυπώσουμε. Τα έχουμε συζητήσει συχνά και είπαμε ότι το Κοινοβούλιο έχει ομοφωνήσει και έχει δεσμευτεί να σας υποστηρίξει σε σχέση και με την νομική βάση ούτως ώστε το ο ESM να αναβαθμιστεί για να πάμε σε κάποιο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με το άρθρο 352 για να δούμε τι εξελίξεις στο Συμβούλιο και στο Eurogroup. Ακόμα δεν έχει επισήμως ε, διαβιβαστεί η πρόταση, το νομικό κείμενο. Τίποτα δεν έχουμε επισήμως λάβει. Ξέρουμε τα κρατημέλη λένε ναι, πρώτα να συζητηθεί το περιεχόμενο και μετά να δούμε το θεσμικό πλαίσιο. Αλλά αυτά πάνε χέρι-χέρι. Επομένως, ήρθε η ώρα να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Ε, είναι κάτι χειροπιαστό αυτές οι εξελίξεις τι είναι, μία φενάκι. Και το έχουμε πει και στο παρελθόν. Τα κράτη-μέλη θα χρηματοδοτήσουν. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία Πολύ σημαντικό αυτό και από θεσμική πλευρά και από πλευρά δυνατοτήτων του. Πώς δηλαδή θα ωφελεί το να γίνει αυτός ο καινούργιο φορέας κομμάτι της θεσμικής αρχιτεκτονικής να βοηθήσει στην σταθεροποίηση γιατί αλλιώς πάνε χαμένα όλα αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να συμβαδίζουν οι αρμοδιότητες οι νέες με τα όσα σήμερα προβλέπονται για πολιτική συνοχή κλπ. Αλλιώς θα είναι θνησιγενές. Άρα είμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική καμπή και θα πρέπει να μας μιλήσουν περί αυτών οι επίτροποι. Τέλος πάντων ήδη φλιάρισα πολύ και ήρθε να σας δώσω τον λόγο. Πρώτα πρώτα, κύριε Ντομπρόφσκης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας ε, και την ακρόαση αυτή ε, από την έκθεση των πέντε Προεδρών και το έγγραφο της Κομισιόν για την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Είχαμε αρκετά εκτεταμένες συζητήσεις και εδώ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με βάση αυτές τις συζητήσεις παρουσιάσαμε ένα πακέτο προτάσεων πέρσι τον Δεκέμβριο. Οπότε είναι χαρά μου που σας ξαναβρίσκω σήμερα. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά ένας τρόπος να επιτύχουμε θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική σταθερότητα. Και οι βασικές αρχές για την Κομισιόν είναι σαφές ενότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Και ε, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η ΟΝΕ και η ολοκληρωσή της πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τους ε, πόρους, ε, ευθύνη και αλληλεγγύη, μείωση του κινδύνου και διαμερισμός του κινδύνου πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι και χρειάζεται μεγαλύτερη συνευθύνη και διαφάνεια και διάλογος με τα Εθνικά Κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους. Μιλώντας λοιπόν για την οικονομική πτυχή του πακέτου μας, η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξή της εδώ και μία δεκαετία, οι επενδύσεις αυξάνεται, η απασχόληση είναι σε επίπεδα ρεκόρ, το επίπεδο ανεργίας είναι σχεδόν σε αυτά προκρίσεις, τα δημόσια οικονομικά βελτιώνονται και ο τραπεζικός τομέας είναι πιο καλά κεφαλαιοποιημένος. Χρειάζεται λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το θετικό περιβάλλον για να ενισχύσουμε τα οικονομικά μας θεμέλια, να σχηματίσουμε κάποια αποθεματικά, να βελτιώσουμε την αντοχή μας και την σύγκληση. Αυτό σημαίνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ολοκλήρωση της τραπεζικής αγοράς και τη αγοράς των κεφαλαιαγορών. Έτσι λοιπόν θα δημιουργήσουμε μια ισχυρή ονέ η οποία θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευημερία. Από τον Δεκέμβριο του 2011 είχαμε πρόοδο στις συστάσεις αναχώρα, οπότε το θέμα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιες χώρες να τα πάνε καλύτερα. Και η Κομισιόν προτείνει να δημιουργήσουμε επιπλέον κίνητρα για τα κράτη-μέλη για να προχωρήσουν σε πολιετήσεις μεταρρυθμίσεις που θα συμφωνήσουν με την Κομισιόν. νομοθετική μας πρόταση θα έρθει τον Μάιο, αλλά η προσέγγιση αυτή ήδη θα μπορούσε να δοκιμαστεί σε μια πιλωτική βάση με το να δοθεί μια επιλογή στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να λύσουν κονδύλια από τα αποθεματικά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών ε, Ταμείων. Γνωρίζουμε ότι αυτό βεβαίως ε, Πρόσκολη σε κάποιε αντιρρήσει, ειδικά την Επιτροπή Ρέτζη, όσον αφορά την πηγή τη χρηματοδότηση, αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει το θέμα αυτό. Δεύτερον, προτείνουμε να αυξηθεί ο προπολογισμό του προγράμματο στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πρόθεσμα μέχρι το 2020, ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τεχνική αρρωγή στα κράτη-μέλη για να προωθήσουν τις ε, μεταρρυθμίσεις. Η συζήτηση είναι αυξημένη, μάλιστα ο προπολογισμό του 2018 ικανοποίησε μόλις το 1 πέμπτο των ετοιμάτων από τα 24 κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θεωρώ ότι το ευρώ για να ευμηνήσει πρέπει να είναι ανοιχτό. Είδαμε στο παρελθόν πως ε, η ολοκλήρωση οδήγησε στην σύγκληση, οπότε θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν στο ευρώ. Και η Κομισιόν ε, προτείνει ότι κατόπιν ετήματος ε, θα μπορούσε να στηρίξει μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν τις χώρες που θα ενταχθούν. Βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μετά το 2020 προτείνουμε ένα ειδικό μέσο σύγκλησης και θα φέρουμε την πρόταση τον Μάιο. Όμως τα μεγάλα σοκ δεν μπορούν ποτέ να αποκλειστούν. Οπότε απαιτείται κάποια εργαλεία για την διαχείριση των κρίσεων Όσον αφορά λοιπόν την άμεση προτεραιότητα μα είναι ακριβώς το να αυξήσουμε το διαμερισμό των κινδύνων και χρειάζεται να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και να υπάρξει μια πραγματική ένωση κεφαλαίου αγορών για την Τραπεζική Ένωση. Τα άμεσα βήματα τα βλέπετε ήδη μπροστά σας και βασιζόμαστε σε εσάς και στους ηγητές ε, Πέτερ Σίμονες, Τερντελάνκε και Χακμαρκ για να ε, καθορίσουν την στάση του Κοινοβουλίου και για το τραπεζικό πακέτο και για το σύστημα εγγύησης ε, των καταθέσεων. γιατί αλλιώς θα εκτεθούμε σε επόμενη μεγάλη τραπεζική κρίση που θα είναι βλαπτική για όλους και βέβαια οι μεταρρυθμίσεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να βοηθήσουν ακριβώς την μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό μας τομέα. Το να συμφωνήσουμε επίση στα εκκρεμή θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Το πρώτο είναι να συμφωνήσουμε στη θέση του Κοινοβουλίου για το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν και ελπίζουμε να τα καταφέρουν να συμφωνήσουν οι ισχυώδεις ηγητές πριν από το καλοκαίρι. Η πρόοδος ε, στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή επίσης έχει σημασία και αναμένουμε και τις σχετικές συμβιβαστικέ προτάσεις. Αλλά οι αγορές ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι από μόνες τους θα εξομαλύνουν ε, τους μεγάλους καράδασμού. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται και ένας δανειστής ε, τελευταίας ε, καταφυγής. Γι' αυτό ακριβώς ε, πρέπει να βασιστούμε στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, βοηθώντας τις χώρες οι οποίες κινδυνεύουν να έχουν χρόνο για να ανακάψουν. Με το να μεταμορφώσουμε το Μηχανισμό Σταθερότητας σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα έχουμε και μεγαλύτερη δημοκρατική εποπτεία και θα μπορούσε ακριβώς να αποτελέσει την δεκλίδα ασφαλείας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Διασώσεων ε, Τραπεζών και για τις, ε, τους μεγάλους ασύμετρους κραδασμούς προετοιμάζουμε μια πρόταση για μια λειτουργία σταθεροποίησης της Ευρωζώνης. Οι εθνικοί υπερπολογισμοί παραμένουν το βασικό μέσο για τις ε, δημοσιονομικές προσαρμογές, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κρατασμοί αυτοί μειώνουν δραστικά το περιθώριο που υπάρχει και γνωρίζουμε ότι ε, συχνά οι επενδύσεις είναι οι πρώτες οι οποίες επηρεάζονται. Οπότε, ως ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Επενδύσεων, ε, κάναμε κάποιες προτάσεις τον Δεκέμβριο, τις οποίες τώρα συγκεκριμενοποιούμε ε, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί βέβαια ένα μηχανισμό μόνιμων μεταφορών κονδυλίων και θα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητα. Τέλο, ε, θέλουμε η ουσία της ε, συνθήκης σταθερότητα και συνεργασία να ενσωματωθεί στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς τα δημοσιοοικονομικά έχουν μεγάλη σημασία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το τρέχον οικονομικό περιβάλλον μας δίνει την δυνατότητα να οικοδομήσουμε μια ανθούσα οικονομία που θα βασίζεται σε γερά θεμέλια για το κοινό μας μέλλον. Έχουμε ένα ολόκληρο έτος να αναμοθετήσουμε πριν τις ευρωεκλογέ και θα πρέπει να το εμμεταλλευτούμε πλήρως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μοσκοσή. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Βάλτης. Όσον αφορά την συνάντηση που λέμε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα για την εμβάνθηση της ε, ΟΝΕ, γνωρίζουμε όλοι ποιες είναι οι πολιτικές και οι οικονομικές ε, προϋποθέσεις στις οποίες εργαζόμαστε, αλλά εννοείται ότι από σήμερα μέχρι τον ε, Ιούνιο θα συνεχίσουμε και θα εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας και δεν πρόκειται να κινηθούμε με αυτόματο πιλότο. Υπάρχει σειρά ε, βημάτων για ανταλλαγή απόψεων, ε, workshop, συνεδριάσεις και την ίδια ώρα όσον αφορά την δέσμη μέτρων που θέλουμε να υιοθετήσουμε Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό που αναφέρατε όσον αφορά το πακέτο μέτρων το προηγούμενο Δεκεμβρίου. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται λοιπόν να μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να υιοθετηθούν και θα πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε σαν ο πυροσβέστης, ο οποίος τρέχει με τον πυροσβεστήρα ενώ έχει ήδη ανάψει η ε, πυρκαγιά. Δεν θέλω εδώ να μειώσω τον ρόλο των πυροσβεστών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να έχει μια προληπτική ε, πολιτική, και ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να συνεισφέρουν και να επωφεληθούν την ίδια ώρα. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και στον τομέα της παιδείας, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε ε, όλους στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Κοινωνική, μια κοινωνία στην Ευρώπη χωρίς ε, αποκλεισμούς. Επίσης, εγώ είμαι πεπισμένος ότι είναι απαραίτητο αυτό που κάνουμε για να συνεχίσουν να υπάρχουν ικανές επενδύσεις σε περίπτωση ασημετρικών σοκ. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ο μηχανισμός σταθεροποίησης θα πρέπει να είναι αξιόπιστος, οικονομικά ισχυρός, έτσι ώστε να μπορέσει να παίξει ένα πραγματικό ρόλο σταθεροποίησης με ικανά κονδύλια και μέσα. Εξού και η πρόταση της Επιτροπής και ξέρετε ότι και για την περιοχή περίοδο συγγνώμη, του πολυμερούς δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020 και όπως ξέρετε εγώ είμαι υπέρμαχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και δεν θα αλλάξω γνώμη τώρα. Στηριζόμαστε λοιπόν στις ίδιες αρχές ισορροπίας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Δημοκρατική ευθύνη και κατανομή του ρίσκου των κινδύνων. Σε αυτό λοιπόν το δημοκρατικό, αν θέλετε, τμήμα της προσπάθειάς μας, τη δημοκρατική της πτυχή, θα ήθελα να πω κάτι εδώ μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημειώνω ότι αυτή η δημοκρατική διάσταση δεν είναι αυτή που βρίσκεται στο προσκήνιο των συζητήσεων μεταξύ κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν πρέπει να την θυσιάσουμε. Δεν πρέπει να την αγνοήσουμε και να την ξεχάσουμε αυτή τη δημοκρατική πτυχή. Και γι' αυτό και θέλω να αναφέρω τρία σημεία. Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης και να ενσωματωθεί αυτός στην νομική τάξη και στο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει εδώ να υπάρξει σημαντική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να ε, αποδυναμώσουμε τα εθνικά κοινοβούλια. Πιστεύω πραγματικά ότι η διακυβερνητική συνεργασία φυσικά είναι κάτι της οποίας ο ρόλος θα πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα στο θεσμικό πλαίσιο και στο θεσμικό περιβάλλον της Ευρώπης η ενσωμάτωση της ε, Δημοσιονομικής Συμφωνίας ε, όσον αφορά την διακυβερνητική της διάσταση είναι κάτι που βεβαίως ενσωματώνεται στο πακέτο μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, μας αφορά η ενίσχυση της δημοκρατικής ευθύνης λογοδοσίας. Και πιστεύω ότι εδώ οι σημαντικές μας προτάσεις θα πρέπει εν ευθέτω χρόνο να δημιουργήσουν νέες αρμοδιότητες για τον πρόεδρο του Eurogroup και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά και νομοθετικά και νομισματικά συγγνώμη, ε, θέματα της Ευρώπης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνεχίζει αυτή η έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και μην ξεχνάμε, γι' αυτό το επαναλαμβάνω στο τέλος της ομιλίας μου, αυτήν την δημοκρατική πτυχή. Μην ξεχνάμε ότι η οικονομική κατάσταση είναι αυτή που είναι, η αποφασιστικότητα των κρατών μελών και ιδιαίτερα της Γαλλίας και της Γερμανίας συνεχίζουν να μας δίνουν ευκαιρίες να προοδεύσουμε και να ξαναδούμε το μέλλον της ε, Οικονομικής και νομοσματικής μας Ένωσης. Ανοίγει ένα παράθυρο, μια ευκαιρία, την οποία δεν πρέπει να γνωρίσουμε, δεν πρέπει να τη χάσουμε. Οι αποφάσεις του Ιουνίου είναι καθοριστικές. Μετά τον Ιούνιο θα είναι πολύ αργά. Σήμερα είμαστε 27 Μαρτίου και μιλάμε για τον Ιούνιο. Λίγες βδομάδες μας μένουν έτσι ώστε το μέλλον της Ευρωζώνης να μπορέσει να αποτελέσει το πραγματικό αντικείμενο αυτής της συνάντησης κορυφής του Ιουνιού. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, όπως σας είπα και σας επαναλαμβάνω και πραγματικά κάνω έκκληση προς όλους σας, ε, προσβλέπουμε και στη δική σας υποστήριξη για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάλτζεκ το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την σημερινή σας ε, παρουσίαση για το πακέτο αυτό από τον Δεκέμβριο ε, το οποίο μας παρουσιάσατε σήμερα είναι οπωσδήποτε πολύπλευρο και η δημόσια συζήτηση δείχνει ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη συζήτησης και ακούγοντας τους κυρίους Ντομπρόφσκης και μοσκόβηση, τότε είναι ακόμη πιο σαφές ότι εντός της Κομισιόν υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση αποκόμισα εγώ. Θα ήθελα να περιοριστώ σε κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα η καλή οικονομική κατάσταση. Αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε, θα έλεγα, σε μία περίοδο οικονομικής επιτυχίας που διορθώνονται οι προβλέψεις ανάπτυξης της Κομισιόν προς τα πάνω και ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή βρίσκεται θα έλεγα περισσότερο στον πολιτικό παρά στον οικονομικό τομέα. Κατά την άποψή μου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εποχή αυτή των παχιών αγελάδων για να δημιουργήσουμε κάποια αποθεματικά και να κάνουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν πιο ανταγωνιστική την οικονομία μακροπρόθεσμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα διαρκήσει αυτή η φάση για πάντα και σε κάποιες χώρες ε, ήδη τα επιτόκια αυξάνονται όπως τις είπα και στην Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν την συγκυρία για να γίνει τώρα πιο ανταγωνιστική η Ευρωζώνη και όλα τα κράτη-μέλη να πατάνε γερά στα πόδια τους για να αντέξουν σε μια ενδεχόμενη κρίση. Οπότε, ποιες είναι οι προτάσεις της Κομισιόν για να υποστηριχθούν οι απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις. Κατόπιν ένα ερώτημα για την σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Έχουμε και ένα πακέτο της ΟΝΕ το οποίο αναφέρατε στο θεσμικό μέτωπο. Βεβαίως, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει η μορφή να ακολουθήσει τους στόχους που έχουμε, να δούμε δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε και μετά να συζητήσουμε τι μορφή θα έχουν. Γιατί οι τίτλοι και τα θεσμικά όργανα σε τελική ανάλυση είναι μόνο θόρυβος εάν δεν συμφωνήσουμε σε κάποιες βασικές αρχές όλοι. και θα πρέπει ακριβώς να υπάρχει εδώ πέρα ένα αίσθημα ευθύνης. Αφού περιγραφούν οι στόχοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Εδώ πέρα λοιπόν θεωρούμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ενισχύσει την πραγματική σύγκληση μεταξύ των ε, κρατών μελών και να δούμε ακριβώς ε, πόσο διατεθειμένα είναι τα κράτη να εφαρμόσουν τις συστάσεις ε, που γίνονται και να ενισχυθούν τα εθνικά κοινοβούλια για να αγκαλιάσουν περισσότερο αυτήν την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. να έρθω πρώτα στο πρώτο σημείο που θέσατε να τονίσω ότι δεν υπάρχουν σήμερα, δεν υπάρχουν διχογνωμίες εντός της Κομισιόν. Οι προτάσεις είναι κοινέ. Ε, τις παρουσιάσαμε από κοινού με τον Επιτροπή Μοσκοβισή και τον Μάιο είναι... Ναι, Ακριβώ θα έχουμε προτάσεις που θα παρουσιάσουμε από κοινού, τις οποίες ε, συζητούμε τώρα εντός της ε, Κομισιόν. Έχουμε μια ομάδα που αφορά ακριβώς την εμβάθυνση της ΟΝΕ, οπότε πρόκειται για ένα αποτέλεσμα κοινή εργασίας. Πρέπει να είμαστε σαφεί. Κατόπιν, για τα ερωτήματα τα οποία θέσατε για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και το ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την αντοχή οικονομιών μας. Αυτό περιέχεται στις ε, προτάσεις μας. Ε, για να παρουσιάσουμε ακριβώς ε, κάποιες προτάσεις Πρώτα απ' όλα, ακριβώς να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κρατών μελών. Δεύτερον, την δυνατότητα και τα μέσα απορρόφησης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όταν ε, θα έρθουν μεγάλοι κράτασμοί και τρίτον να διευκολύνουμε την σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Και ακολουθούμε και τα τρία αυτά παράλληλα και θα έλεγα ότι συμφωνώ με αυτό. Ναι, ναι πρόκειται για συλλογικό χαρακτήρα που έχουν οι προτάσεις όπως είπε ο συνάδελφος. Είναι ομαδική η δουλειά μας. Βρίσκεται σε αυτές τις προτάσεις όλη η Επιτροπή. Σωστά το είπε ο κύριος Μπάλτσα. Είναι πιο ενάρετος τώρα ο οικονομικός κύκλος. Όχι όμως, θα εντύρουμε τις προσπαθειές μας, παρά αυτά, ούτε πρέπει να αγνοήσουμε τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κάποιων κρατών μέλων. και της Ευρωζώνης. Είπαμε για τα κόκκινα δάνεια που είναι κοινό πρόβλημα, μειώθηκαν πάντως και όσον αφορά την ε, Τραπεζική Ένωση, έχουμε τον εποπτικό μηχανισμό, όλα αυτά δεν τα είχαμε επικρίσεως. Και γι' αυτό σας λέω. Το backstop, ε, η Τραπεζική Ένωση, όλα αυτά είναι η εμβάθυνση της Νομισματικής Ένωσης. Μπέρε, σας ευχαριστώ. Θεωρώ θετικά το όσα ακούσαμε σήμερα για τα μέτρα του Δεκεμβρίου. Κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόσκης, μας ε, αναφέρατε πάλι τη πρόοδος που σημειώνεται για την Τραπεζική Ένωση και για τις κεφαλαίες και πρόκειται για δύο μέτωπα πολύ σημαντικά. είναι θέμα της εμβάθμισης της νομισματικής ένωσης. Και υπάρχουν διάφορες προτάσεις, διάφορες ιδέες που κυκλοφορούν και άρα θα πρέπει να διορθώσουμε τη ρότα που έχουμε πάρει σχετικά με αυτά και σε σχέση με την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο για το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μοσκοβισή την περασμένη εβδομάδα. Είναι σημαντικές κάποιες βασικές αρχές. Πέραν του, της υπόθεσης του ονόματος, τελείωσε αυτή η υπόθεση. Τώρα έχουμε κάποιες καθεντήριες γραμμές που πρόκειται να ζητηθούν στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να προσέξουμε μόνο στα εξή. Πρώτα-πρώτα, το άρθρο 4 του Νομισματικού Ταμείου δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στα του Ευρωπαϊκού Ταμείου όσον αφορά την νομική πειθαρχία. Επίσης, στην νομοθεσία μας έχουμε κάποιες ε, ασφαλιστικές δικλείδες. Έχουμε δημοκρατικό πλαίσιο, άρα δεν ε, έχει νόημα η αναπαραγωγή των όσων ισχύουν στο δούνο του. Ε, αυτά λένε τα εφαρμόσουμε όχι ε, όχι όσα ισχύουν στην λεγόμενη Τρόικα. Αλλά πρέπει να υπάρχει προβληματισμό όσον αφορά το aggregate fiscal stand. Και να προετοιμάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις της χρονιάς. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όσον αφορά το δημοσιονομικό σύμφωνο, νομίζω ότι έχετε αναθέσει στην νομική σας υπηρεσία να δείτε κατά πόσον ε, αυτά συνάδουν προ το six pack, το two pack και εν συνάδω προς τη διαδικασία της συναπόφαση. Πάντως, το Μάιο περιμένω την πρότασή σας για τη λειτουργία της σταθεροποίησης. Και να δούμε αν θα συμφωνήσουν οι τεχνοκράτες με τους πανεπιστημιακούς. Άρα, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προτάσεις που να συνάδουν με τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Και στην πολιτική μας ομάδα η οικογένεια θα πρέπει κάτι να κάνουμε για την αντιμετώπιση της ανεργίας και έτσι να προχωρήσουμε στην εμβάθυνση της Νομισματικής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέρες, λέει ο κ. Μοσκοβίζη, σωστά υπενθυμίσατε ότι το θέμα είναι ακόμα ανοιχτό. Πρώτος έχουμε συζητήσει για την εμβάθυνση της Νομισματικής Ένωσης. Πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πώς το νόμισμά μας θα είναι εγγύηση σταθερότητας. Πώς θα έχει οικονομία δυναμικό χαρακτήρα, θα ενθαρρύνονται οι επενδύσεις, και θα πρέπει να ξεχνάμε τη δημοκρατική διάσταση του πλαισίου μας. Συνεργαζόμαστε με το Fiscal Board. Ακολουθούμε τις προτάσεις του. Αλλά δεν χαλαρώνουμε την στήριξη της οικονομίας και για την σταθεροποίηση λαμβάνω υπόψη αυτά τα οποία είπατε για την συνέχεια της προβληματικής μας. Ντομπρόσκης, όχι. Ναι, πείτε προς Ντομπρόσκης. Να συμπληρώσω σε αυτά που ακούσαμε. Πρώτο πρώτο αυτό που είπατε για την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των αγορών αυτά δεν υποκαθιστούν την ε, εμβάθυνση της νομισματικής ένωσης. Πρόκειται για προτεραιότητες. Η τραπεζική μεταρρύθμιση του Νοεμβρίου του 2016 ελπίζουμε να εγκριθεί του αμέσως επόμενους μήνες από το Συμβούλιο. Και έχουμε και τη φάση του τριμερούς διαλόγου. Οπότε να υπάρξει συμφωνία επί της αρχής και για τα το το για το Συμβούλιο Εξυγίανσης και έχουμε υποβάλει νομοθετικές προτάσεις από τις οποίες έχουν εγκριθεί μόνο τρεις. Άρα ακόμα υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει και δουλειά σημαντική. Πάντως αυτά τα δύο μέτωπα, παραβάνω είναι συμπληρωματικά και δεν αλληλοανερώνται. Πρώτος, Γουαλθιέρη. βεβαίω και εμείς είπαμε ότι θα πρέπει ταχαίως για το backstop, για όλα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουμε και για το NPL, για τα δάνεια να προχωρήσουμε ταχαίως. Τέλος πάντων, όσον αφορά το θέμα της ονομασίας που ανέφερε η Περβάνος Μπερές, ότι το, το, όνομα είναι απόρρια της ουσίας του πράγματος στα λατινικά. Αλλά να, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Γιατί εδώ πέρα πρόκειται για κάποια εξαιρετικού χαρακτήρα ρύθμιση. Οπότε λέμε, μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ε, Επόμενο ομιλητή. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και κάποιος καθηγητής ανέφερε το ότι υπάρχουν πολιτικοί και τεχνοκρατικοί λόγοι γιατί πρέπει να συγκροτηθεί ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, νομισματικό ταμείο. Δεν είναι πολιτικοί λόγοι. Γιατί ε, πρόκειται τώρα για αναπτυγμένες χώρες από την άλλη μεριά Οι πόροι του Δουνουτού δεν αρκούν να σώσουν κάποια χώρα. Τα προβλήματα της χρηματοοικονομικής κρίσης ακόμα υπάρχουν. Α, είδατε, είχαμε επίσης σχέση με την κρίση στην Ελλάδα, να σταθεροποιήσουν τις αγορές, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει ε, να βοηθούν οι χώρες να σταθεροποιηθούν. και θα πρέπει να δημιουργηθούν ευμενείς οικονομικές συνθήκες και να διορθωθούν τα λάθη που έχουν γίνει. Μα υπάρχουν οικονομικοί λόγοι για τους οποίους θα προχωρήσουμε προς το Ευρωπαϊκό Μεσματικό Ταμείο, μα έχουμε το ΔΝΤ, το οποίο ήδη ε, σχετίζεται με τόσες κρίσεις. Well, uh, on the question on, uh, uh, για το θέμα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να σας πω ότι ήδη ε, μάθαμε στην κρίση της ε, Ευρωζώνης ε, πως χρειάζεται ένας μηχανισμός εκτακτής στήριξης για τα μέλη της Ευρωζώνης και υπήρχε μια, ένα ειδικό μέσο ε, για την Ελλάδα, υπήρχε ο μηχανισμός EFSF και τελικά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας που δημιουργήθηκε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δίδαγμα και μια εμπειρία από την κρίση ότι χρειαζόμαστε έναν τέτοιο μηχανισμό ε, ακριβώ επειδή υπάρχουν και όρια στο σε ποιο βαθμό είναι το ΔΕΛΤΕΝΤΑΦ διατεθειμένο να εμπλακεί σε προγράμματα στην Ευρωζώνη και σε χώρες της Ευρώπης ε, ως ε, ανεπτυγμένες οικονομίες ε, θα πρέπει να μπορούμε να φροντίσουμε αυτούς. Οπότε ο ρόλος μας υπάρχει, αλλά η τωρινή συνθήκη του Μηχανισμού Σταθερότητας λέει ότι τα προγράμματα αυτά γίνονται από την Κομισιόν ε, σε στενή συνεργασία με το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, αλλά όπως βλέπετε στο τελευταίο ελληνικό πρόγραμμα, το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ ε, δεν συνεισφέρει οικονομικά, οπότε αυτό είναι ένα μήνυμα ότι χρειάζεται ένας ισχυρότερος ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ε, πιθανώς προς ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε και οι δύο τονίσατε πόσο σημαντικό είναι να γίνει ο μηχανισμός σταθερότητας ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Και είπατε πως ε, αυτά θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Εγώ βλέπω πως ε, λίγα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να αποκλίνουν από τη διακυβερνητική μέθοδο και ε, βλέπουμε, την, και βλέπουμε ότι αυτό προτιμάται τελικά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε διακυβερνητικέ ε, συνεννοήσεις και όχι κοινοτική μεθόδο. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που δεν περάσει λοιπόν κάτι τέτοιο στο Συμβούλιο. Εσεί, κύριε Μοσκοβισή, είπατε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο εμπόδιο. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Δεύτερη ερώτηση για τον λεγόμενο Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, ξεκαθαρίσει πως ε, δεν θεωρούν την Κομισιόν κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέση λοιπόν θα έχει αυτός ο Υπουργός Οικονομικών, θα είναι επικεφαλής της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα θα έχει και άλλη λειτουργία, ε, αρμοδιότητα εκτός Κομισιόν ή θα είναι σαν την κυρία Μογκερίνη μέλος της Κομισιόν και ταυτόχρονα κεφαλή της Ευρωζώνης. Ε, στην περίπτωση αυτή ο Υπουργό Οικονομικών, το λέει και το όνομα άλλωστε, θα έχει ε, έναν ρόλο κυβέρνηση κάτι το οποίο απορρίπτουν οι εθνικές ε, κυβερνήσει. Τι θα κάνετε με αυτό το δίλημα. Και τέλος ε, έχουμε την μεγάλη, για να μην πω υπερβολική αμοιβαία εξάρτηση των κυβερνήσεων και των κρατών, των τραπεζών και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Δηλαδή, Αναφέρομαι στα κρατικά ομόλογα τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν χωρίς να διαθέσουν κεφάλαια οι τράπεζες. Πώς σκοπεύετε να ξεπεράσετε αυτή την αμοιβαία εξάρτηση για να διασφαλίσετε ότι στο μέλλον οι τράπεζες δεν θα διατρέχουν αυτόν τον σωρευτικό κίνδυνο. Λοιπόν, για τις τρεις αυτές ερωτήσεις. Η πρώτη για την κοινοτική μέθοδο σε αντίθεση με την διακυβερνητική. Πρέπει να πούμε ότι ήδη όταν φτιαχνόταν αυτοί οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είχε τότε ήδη συμφωνηθεί ότι ε, για λόγους ε, ταχύτητας και πρακτικότητας ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης θα γίνουν τα πράγματα διακυβερνητικά, αλλά θα πρέπει τελικά να ακολουθηθεί η κοινοτική μέθοδος. Αυτό είχε συμφωνηθεί ήδη αρχικά στην περίπτωση της σχετικής συνθήκης υπήρχαν και συγκεκριμένες προθεσμίες. Οπότε, τι κάνουμε εδώ πέρα. Ακολουθούμε τις ε, αρχικές ε, συμφωνίες ε, και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας προτείνουμε και κάποιες νέες αρμοδιότητες όπως την διασφάλιση για ένα ευρωπαϊκό ενιαίο Ταμείο Διάσωσης και μία δημοσιονομική λειτουργία της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η πρότασή μας. Τώρα βεβαίω είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με τα κρατημέλη, με το Κοινοβούλιο, να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή την προσέγγιση και προφανώς ως Κομισιόν ε, υπερασπιζόμαστε την κοινοτική μέθοδο. Κατόπιν για το θέμα του Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών. Αυτή είναι μια πρόταση η πρόθεσμη. Η ιδέα αυτής της ε, διπλής δομής θα ήταν, ε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πράγματι ε, κάτι πιο κοντά στο πώς λειτουργεί η πατή εκπρόσωπος, δηλαδή θα είναι πρόεδρος της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα μέλος της Κομισιόν αρμόδιο για την ΟΝΕ να έχει λοιπόν αυτά τα δύο χαρτοφυλάκια. Και πράγματι την έμπνευση την αντλήσαμε από αυτό το οποίο ισχύει ήδη ε, στα εξωτερικά. Και κατόπιν ε, για τον δεσμό τραπεζών και κρατών που αναφέρατε, μια άμεση πρόταση που θα υποβάλουμε προσεχώς είναι να τοποθετηθεί και να είναι αρμόδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας για τα ζητήματα κρατικών ομολόγων ακριβώς δηλαδή για το δημόσιο χρέος της ε, Ευρωζώνης ε, και τα σχετικά ομόλογα και στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες να μην εκτίθενται τόσο πολύ στο οικείο κράτος αλλά να μπορούν να έχουν ένα πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Και βεβαίως προσεχώς ακριβώς θα προχωρήσουμε σε, μηδεν... σε εξελόγηση μηδενικού κινδύνου για τα ομόλογα που είναι μια προϋπόθεση για να συμβεί αυτό. Μετά υπάρχει μια ξεχωριστή συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζονται ρυθμιστικά οι εκθέσεις, ε, τα ανοίγματα σε ξένα ε, κράτη. Εδώ οι απόψεις ε, διήστανται. Ε, γνωρίζουμε ότι τον Ιούνιο του 2016 είχαμε συμφωνήσει να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο γίνεται στην Βασιλεία σε διεθνές επίπεδο. Έχει ολοκληρωθεί όμως, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην Βασιλεία χωρίς να καταλήξουν κάπου, οπότε δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με προσοχή γιατί μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες για την δημοσιονομική σταθερότητα των κρατών μελών εάν βιαστούμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ. Δύο λόγια μόνο θέλω να προσθέσω. Εγώ βεβαίως πιστεύω ότι η πιο δημοκρατική μέθοδος είναι η κοινοτική μέθοδος, αυτή που επιτρέπει τον δημοκρατικό έλεγχο. Χωρίς ε, δημοκρατική διαδικασία και δημοκρατικό έλεγχο, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι για το μηχανισμό σταθερότητας αυτό θα πρέπει να ισχύσει. Καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις των κρατών μελών Χρειάζεται όμως μία εξέλιξη μέσω πρόθεσμα και ξέρω ότι στη Γερμανία η διακρατική συμφωνία προς τα εκεί πάει. Ενισχύεται λοιπόν αυτή η υπόθεση εργασίας όλο και περισσότερο. Ένας υπουργό ε, υπουργός για την Ευρωζώνη με ένα ρόλο παρόμοιο με αυτό της κυρίας Μογκερίνη σήμερα σαφώς και είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε τον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου σήμερα. Και για μένα όσο πιο γρήγορα γίνει κάτι τέτοιο και υλοποιηθεί αυτή η ιδέα τόσο το καλύτερο. Και νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον χρόνο για χάσιμο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, επαναλαμβάνω, δεν είναι η άποψη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Αντιπρόεδρε, θυμάμαι τι είχατε πει για το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας την προηγούμενη φορά. Αναφερθήκατε στις διάφορες χώρες στη σχέση με τις τράπεζες, και ουσιαστικά τους κανόνες μας που τους υποχρεώνουν να αντιμετωπίσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα επικίνδυνα στοιχεία του ενεργητικού. Η κυρία Μιράντα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εννοείται ότι το πακέτο αυτό είναι μια χαμένη ευκαιρία υπάρχουν αδυναμίες και εμείς ε, ουσιαστικά προχωρούμε με πάρα πολύ διστεκτικά βήματα για να καλύψουμε αυτή την έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο για μας έχει ανύπαρκτο ελεγκτικό και εποπτικό ρόλο. Και το δίκτυο προστασίας... Αλλά και για μένα και για τον συνάδελφο Ουρτάσου που έχουμε περάσει στην Ισπανία διαρθρωτικές πολύ σκληρές μεταρρυθμίσεις εις βάρος του Κοσμάκη και έφεραν φτώχεια, έφεραν κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, ε, ε, αυτό το πακέτο σφραγίζει τις χρυσούς κανόνες που αφορούν την λιτότητα. Άρα δημοκρατικά θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσης, για πέστε μας, κάντε μας μια αξιολόγηση όσον αφορά το πρόγραμμα στήριξης των διορθωτικών μεταρρυθμίσεων. Αντιπρόεδρε, επίτροπε, δεν αμφιβάλλουμε ως κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε κατά των προϋποθέσεων για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Τα είπαμε και στην ε, Ολομέλεια είχαμε απευθύνει ερωτήσει περιβαλλικής πολιτικής προς την Επιτροπή και είναι κρυστάλλινη η θέση μας σε σχέση με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Θεωρούμε ότι αυτά αποτελούν ράπισμα για όλους όσους είναι δικαιούχοι των διορθωτικών πόρων. Δεν γελιόμαστε γι' αυτά. Και στους δύο απευθύνεται αυτή η ερώτηση. Πρόκειται να εγγυηθείτε το ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα οδηγήσει σε επιδείνωση των κοινοφελών υπηρεσιών και σε ιδιωτικοποίηση. Είναι ελάχιστα δημοφιλή αυτά τα μέτρα στα κράτη-μέλη. πρόκειται αυτά τα μέτρα να περάσουν από τα εθνικά κοινοβούλια. Πώς έτσι θα εγγυηθείτε την δημοκρατική νομιμότητα και κάποια συνένεση για αυτές τις μεταρρυθμίσει μεταρρυθμίσεις επίσης και πώς θα συμμετάσχουν κατά κάποιο τρόπο οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτά. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Βουλευτή ότι η Επιτροπή αυτή στηρίζεται σε κανόνες και φυσικά Θέλουμε να μειώσουμε το έλλειμμα και να υπάρχει μια δημοσιονομική πειθαρχία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της λιτότητας, της δημοσιονομικής λιτότητας σαν Επιτροπή. Και μέσω της τάσης μας, και αυτό το δείξαμε στην ελληνική κρίση, θέλουμε να επιλεγεί η δημοσιονομική σοβαρότητα με φυσικά την ανάπτυξη. Και σε κάθε περίπτωση ε, θέλουμε κάποια ευελιξία δημοσιονομική. Σήμερα είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντική μείωση λοιπόν των ελλημάτων και ελπίζω ότι όλες οι χώρες θα βγουν από αυτό το υπερβολικό έλλειμμα στο οποίο βρίσκονται κάποιες. Δεν προτείνουμε λιτότητα, προτείνουμε μηχανισμούς σταθερότητας για να μειωθούν οι διαφορές και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Κύριε Πρόεδρε, εννοείται ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη στρατηγική μας για τη μείωση των διαφορών και την σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός μας δεν είναι η άκρατη ιδιωτικοποίηση, η απορρίθμιση και η κατάργηση των κανόνων. Βρισκόμαστε σε μια οικονομία ψηφιακή όλο και περισσότερο και η μεταρρύθμιση την οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε, μια μεταρρύθμιση η οποία θα πρέπει να εμπλέκει όλους τους τομείς. Την καινοτομία, την έρευνα, και φυσικά την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόεδρος, να συμπληρώσω κάτι. Για τις ε, μεταρρυθμίσεις. Εάν δείτε, παραδείγματος χάρη, το πρόγραμμα στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αυτό βασίζεται στην ζήτηση. Ε, δηλαδή τα κράτη-μέλη ζητούν στήριξη για μεταρρυθμίσεις που καθορίζουν τα ίδια όταν ε, αξιολογούμε αυτά τα αιτήματα λαμβάνουμε υπόψη ε, το εάν ευθυγραμμίζονται με τις ε, συστάσεις αναχώρα το πώς ευθυγραμμίζονται με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, το εάν είναι όντως σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα κριτήρια και όπως σας είπα, βασίζονται στην ζήτηση και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν για ποιες μεταρρυθμίσεις ζητούν στήριξη και παρόμοιο είναι το σκεπτικό όταν προτείνουμε ακριβώ αυτό το εργαλείο για τις μεταρρυθμίσεις ε, όπου τα κράτη-μέλη έχουν οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή κάποιων μεταρρυθμίσεων. Κύριε Παπαδημούλης. Πρόεδρε, επιτρέψτε με να σας ρωτήσω ε, για τη χώρα μου την Ελλάδα. Σημειώνω με ικανοποίηση τις θετικές εκτιμήσεις της Κομισιόν για την πορεία, την επιτυχή της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Σημειώνω όμως επίσης ότι υπάρχει μια δέσμευση και από τις ελληνικές αρχές και από τον ESM και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Κομισιόν για ένα πολύ εντατικό χρονοδιάγραμμα υλοποίηση στόχων έτσι ώστε το αργότερο στις αρχές Ιουλίου, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, αρκετά πριν την τυπική λήξη του προγράμματος, να έχει ολοκληρωθεί όλο το πακέτο των συμφωνημένων βημάτων. Η τέταρτη και τελική αξιολόγηση, το ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 100% ελληνικής ιδιοκτησίας για την περίοδο μετά το τέλος των προγραμμάτων, που αυτά κυρίως βαραίνουν την Ελλάδα ως υποχρέωση επισπεύδοντος, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που κυρίως βαραίνουν το, την πλευρά των δανειστών. Η συγκεκριμενοποίηση των μέτρων ελάφρυσης του χρέους των μεσοπρόθεσμων με βάση όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί ομόφωνα στο Eurogroup στις 15 Ιουνίου του 2017, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των κανόνων εποπτείας της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος του προγράμματος με βάση τον κανονισμό 472 του 2013. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Λίγους μήνες πριν το τέλος του τρίτου προγράμματος, τρία χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα μετάσχει το πρόγραμμα. Και επιπλέον όλοι οι, όλες οι εκτιμήσεις για την πορεία των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, της Κομισιόν, έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Επειδή στο παρελθόν είχαμε καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από ενστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ζημίωσαν την οικονομία της ε, Ελλάδας και το λαό της Ελλάδας. Και επειδή οι καθυστερήσεις είναι επιζήμιες, σας ερωτώ πώς σκοπεύετε να κινηθείτε έτσι ώστε να έχουμε έγκαιρη ολοκλήρωση και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Και ποιος θα είναι ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μετά τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Euh, Για να ολοκληρωθεί εγκαίρως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οι αποφάσεις θα ληφθούν θεωρητικά στις 21 Ιουνίου το Eurogroup, ίσως λίγο αργότερα, εν πάση προθεσμία σήμερα είναι 21 Ιουνίου. Γνωρίζετε ποια είναι αυτά που πρέπει να ολοκληρώσουν οι ελληνικές αρχές, τα γνωρίζετε κύριε Βουλευτά, στρατηγική ανάπτυξης που θα πρέπει να σχεδιαστεί από τους Έλληνες, για τους Έλληνες, που να προσαρμόζεται στα ελληνικά δεδομένα. Πρέπει να υιοθετηθούν κάποια προαπαιτούμενα, νομίζω το Μάιο, και θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και ποια θα είναι η παρακολούθηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση και στο Eurogroup και στο Euro Working Group ε, δεν έχουμε ξεχάσει το μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους. Θα πρέπει να γίνει αυτό σε συνδυασμό με την επιστροφή της ανάπτυξης και βεβαίως το θέμα της παρακολούθησης ε, των ελληνικών τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τους άλλους θεσμούς για να προετοιμάσουμε την έξοδο και φυσικά η αξιολόγηση είναι κάτι καθοριστικό γι' αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι μυστικό ότι υπήρξαν ε, τεχνικές συζητήσεις στο παρελθόν ε, μεταξύ Δουνουτού και Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα στοιχεία και τους αριθμούς και σε γενικές γραμμές μπορώ να σας πω ότι οι αριθμοί και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα και όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και όσον αφορά τα άλλα στοιχεία, η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική πρόοδο. Ελπίζω λοιπόν ότι στη συζήτηση που θα συνεχίσουμε να έχουμε με τους φίλους μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα τους πείσουμε. Ε, το βασικό είναι ότι λαμβάνονται μέτρα, ότι η ανάπτυξη επιστρέφει, βελτιώνει την κατάσταση δεν χρειάζεται κάποιο να έχει βγάλει πανεπιστήμιο μαθηματικών για να καταλάβει προς τα που πρέπει να πάμε. Και φυσικά οι συναντήσεις, ε, οι γενικές συνελεύσεις του Διεθνούς Δομιστικού Ταμείου και όλες οι επαφές που έχουμε μαζί τους θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα είμαστε αντικειμενικοί. Θα είμαστε ειλικρινείς, αντικειμενικοί και απαιτητικοί βεβαίως. Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τους δύο επιτρόπους για τα όσα μας ε, ανέπτυξαν και και όπως όλοι οι συνάδελφοι και όταν τα παρακολούθησα με προσοχή θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί κάποια λύση που να διακρίνεται από οικονομική ισορροπία γιατί η Νότια Ευρώπη δεν μπορεί παρά να θέλει να πιάσουν το προσπάθειές της. Το πρόβλημα είναι ότι οι σημερινοί συμβιβασμοί δεν επιλύουν το πρόβλημα της οικονομικής ανισορροπίας γιατί υπάρχουν κάποια μέσα ε, αυτά τα 20-25 δις ε, για τον προϋπολογισμό έχουν κάνει λοιπόν θυσίες τα, τα κράτη-μέλη εκεί στην Νότια Ευρώπη αλλά διεπονται τώρα από αυτή την φάση της δημοσιονομικής λιτότητας. Άρα χρειάζεται να βρούμε κάποια ισορροπία, να βρούμε κάποια εργαλεία τα οποία να διέπονται από τις εύστοχες προϋποθέσεις. Και η Ιταλία χρειάζεται πόρους. Και να μην έχουμε μεταρρυθμίσεις που να μην είναι δημοφιλής γιατί είναι άδικες. Ξέρω ότι υπάρχει ευαισθησία από πλευράς Επιτροπής, αλλά και το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να θέλει κάποια πράγματα τέτοια όπως αυτές τις δημοσιονομικές ε, ε, αλλαγές. Επομένως, όχι πια συμβασμοί οι οποίοι δεν αποδίδουν το ESB και το ευρωομόλογο θεώρησε, θεωρήθηκε ότι θα μπορέσει να είναι μια λύση και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια δίκη κατανομή των κινδύνων. Θα έχουμε ένα εργαλείο το οποίο να είναι όμως, θα πρέπει να είναι, διαρκής λύση και όχι ένας συμβιβασμός. Να μην οδηγούμεθα σε χρεοκοπία. Θα ξανάρθει η κρίση κυκλική. Και η Ευρωζώνη είναι θωρακισμένη, να μην στερείται των μέσων εξέβρεσης λύσεων. Yeah, uh, um, uh, uh, Σε ευχαριστώ για όσα είπατε, λέει ο κύριος Αντιπρόεδρος Επιτροπής. Τώρα, σε σχέση με το τι θα κάνουμε με τις οικονομικές ανισορροπίες. Ακριβώς προς τα εκεί κατατείνουν οι προτάσεις μας. Οπότε, έχουμε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα πρώτα για το πώς θα θωρακίσουμε την Ευρωζώνη και τις οικονομίες της επίσης, ε, θα, ο άλλος άξονας των πιθουλεύουν πώς θα βελτιώσουμε το μηχανισμό απορρόφησης των κρίσεων. Αυτά, αυτά θα μας απασχολήσουν. Πρώτα πρώτα όσον αφορά την στήριξη των ε, διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και τα μέσα τα οποία θα μετέλθουν τώρα όσον αφορά τα στοιχεία ακόμα δεν έχουν αποκριστελωθεί. Ε, γι' αυτό μιλάμε για discussion paper, ακόμα αυτά τα κουβεντιάζουμε. Αρχάς, Μαΐο σε σχέση με το πολιτές δημοσιογικό πλαίσιο θα τα δούμε όλα αυτά οριστικά. Άρα, θέλουμε έναν μηχανισμό από πλευρά ζήτηση, έτσι να έχουμε κάποια κίνητρα στήριξη των κρατών μελών, ε, δηλαδή να μην έχουμε ε, δάνεια, να έχουμε επιδότηση, να έχουμε ενισχύσει. Τέτοιου είδου χρηματοδότηση να δώσουμε στα κράτη-μέλη για τι μεταρρυθμίσει. Επίση, για τη σταθεροποιητική λειτουργία της Ευρωζώνης. Όντως, βασικά προβλέπονται τα δάνεια ως ε, μέσο, ως εργαλείο. Αυτό όμως είναι για να στηρίξει τις ε, κρατικές επενδύσεις στα κράτη-μέλη όταν έχουμε τα, τα, τα μεγάλα ασυμμετρικά σοκ. Γι' αυτό και εμείς βοηθούμε για τέτοιες επενδύσεις και είπαμε ότι ε, μπορεί, έχουμε βασικά δάνεια και επικουρικά έχουμε και τις ενισχύσεις ε, επιδοτήσεις. Αυτά τα δύο εργαλεία μεταρχόμαστε. Επίσης, για τα ευρωομόλογα έχουν γίνει συζητήσεις και στο παρελθόν. Και ακούσαμε και το τι, τι έχουν να το feedback. και για το EMU. Τα συζητήσαμε. Και σε πρώτη φάση δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα. Θέλουμε κρατικά ομόλογα να χρησιμοποιούνται. Oui, je veux assurer, euh, monsieur... Ναι, κύριε Βουλευτά, η πρόθεση της Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν είναι να παρέμβει στις δημοκρατικές διαδικασίες και μπορείτε βεβαίως να υιοθετήσετε τις μεταρρυθμίσεις που επιλέγετε. Αλλά όλοι ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την πολύ αδύναμη παραγωγικότητα που παρατηρείται στην Ιταλία και εδώ αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επίσης το χρέος της Ιταλίας είναι υψηλό, πρέπει να μειωθεί. Και βεβαίως στηρίζουμε την ανάπτυξη, αλλά χρειάζεται και μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Η μεγάλη χώρα που είναι η Ιταλία, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και πολύ γρήγορα θα είναι και η τρίτη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμευμένη στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, θα πρέπει να εφαρμόσει τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Και αυτό είναι κάτι θετικό, γιατί πολεμά το χρέος, που είναι κάτι που θα επομισθούν οι επόμενες γενιές ο Μπερνάρ Μονό. Κύριε Επίτροπη, μπροστά στην αποτυχία της Ευρωζώνης, η φυγή προ τα μπρο είναι η μόνη λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνεται λοιπόν να εμβαθύνουμε περισσότερο την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή με χύψη πακέτα μέτρων. Για μα βεβαίω αυτό είναι η χειρότερη λύση. Αυτό το έχει αποδείξει και το παρελθόν. Ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνοντας τον έλεγχο των δημοκρατικών ελόφων από τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό το ονομάζετε εσείς ανεξαρτησία. Κατόπιν εδόθη η αρμοδιότητα αυτή στα, στην Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή, κάτι που αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα επιλογής των κρατών μελών. Και το τρίτο στάδιο που προτείνεται είναι η υποταγή. Βλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί ένας Ευρωπαίος χωροφύλακας, ο οποίος θα μπορεί να επιβάλλει μέτρα λιτότητα σε δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, υποσχόμενοι κάποιες μικρές ε, παρεμβάσεις και βοήθεια όταν υπάρξει οικονομική κρίση και αποκλεισμό από τις χρηματαγορές όπως έγινε στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά εδώ καταστρέφεται τα οικονομικά μέσα και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομισματικό Ταμείο δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ε, καταστροφικές συνέπειες. Τα χρέη που πλήττουν τα κράτη-μέλη είναι κάτι το εξαιρετικά βαρύ. Εσείς αναπτύσσετε εργαλεία και μέσα που πραγματικά δεν είναι αποτελεσματικά. Δεν επιτρέπεται στις τράπεζες να χειριστούν τα διεθνή μέσα που διαθέτουν βλέπετε ότι όλα αυτά που κάνετε είναι πολύ χρήσιμα για τις Ηνωμένε Πολιτείες και για την Goldman Sachs. Βλέπετε ποιος πήρε σήμερα την θέση του Υφυπουργού στη Γερμανία υπεύθυνου για την οικονομική πολιτική. Κάποιος που προέρχεται από την Goldman Sachs. Μειώνεται λοιπόν τον δημοκρατικό έλεγχο που θα μπορούσε κάποιος να ασκήσει κατά αυτού του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Ο κύριος Μοσκοβίση. Κύριε Μονό, ακούγοντάς σας κάτι δεν καταλάβαινα. Αρκετά δεν καταλάβαινα. Ίσως είμαι περιορισμένη ευφυΐας. Αλλά και ο τρόπος που εκφράζεστε, αν θέλετε, είναι ασαφής. Δεν καταλαβαίνω. Είστε υπέρ ή κατά του ευρώ. Θέλετε να παραμείνετε στο ευρώ ή να βγείτε από το ευρώ. Μιλάτε για δημοκρατικές επιλογές. Οι δημοκρατικές επιλογές πάντως που έκαναν οι πολίτες της χώρας μας είναι πολύ συγκεκριμένες. Και αν θέλετε η Ευρωζώνη δεν είναι απλώς μια ιδεολογική επιλογή που πολλές φορές μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Οι πολίτες της Ευρώπης δεν κάνουν λάθος παρόλα αυτά. Ξέρουν ότι το ευρώ αποτελεί προστασία. Επιτεθήκατε ως συνήθως θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χωρίς όμως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χωρίς τις επιλογές του Μάριο Ντράγκη το 12, χωρίς τα προγράμματα για την ρευστότητα στην Ευρώπη, δεν θα βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα με εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό και με μια ανάπτυξη για τους περισσότερους. Θα είχαμε spread ανησυχητικά τεράστια, τα οποία θα είχαν οξύνει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Οι μηχανισμοί εποπτείας, οι μηχανισμοί για τα τραπεζικά θέματα, οι οποίοι έχουν σήμερα επικρατήσει. Οι μηχανισμοί για τις πτωχεύσεις μας προστατεύουν. Το ευρώ λοιπόν μην το αγνοείτε, γιατί αυτό είναι ανόητο. Δεν έχει ε, τίποτα άλλο σήμερα στην Ευρώπη από το να προστατεύσει όλα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι κάτι που το προβλέπουν οι συνθήκες και βεβαίως ο τρόπος που αυτό θα γίνει θα περιέχει και στοιχεία ευελιξίας. Αυτό λοιπόν που λέτε, αυτό που σκέφτεστε για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και από την αποστολή σας. Και πιστεύω ότι επικρατεί σύγχυση στο μυαλό σας. Κύριε Επίτροπε, δεν απαντήσατε όμως όσον το δημοκρατικό χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Δημοσιου. Νομισματικού Ταμείου, Μοσκοβισή, η Επιτροπή προτείνει να ενσωματωθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος, κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ο καλύτερος τρόπος να αυξηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και αυτό δεν το καταλάβετε. Τι έχετε να πείτε για τα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και συμφωνώ με τα όσα είπε ο Επιτροπός Μοσκοβισή και επίσης ε, και με την παρατήρηση για την δημοκρατική νομοποίηση η οποία βεβαίως δεν θα πρέπει να θυσιάζεται και επειδή θεωρώ ότι εάν θυσιαστεί ε, δεν θα έχουμε αποτελεσματικότητα και στις άλλες ε, διαστάσεις. Γι' αυτό ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν την πρόταση της ε, Κομισιόν και να ενταχθεί το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο στην κοινοτική μέθοδο και αναμένουμε και μια φιλόδοξη πρόταση για τα υπόλοιπα στοιχεία του πακέτου της ΟΝΕ. Εμείς από την πλευρά μας βεβαίως θα προσπαθήσουμε παράλληλα να ολοκληρώσουμε τους νομοθετικούς ε, φακέλους. Ε, υπάρχει ακριβώς ε, και ένας καταμερισμός του κινδύνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε οπωσδήποτε τον διάλογό μας. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Διάλειμμα ενός λεπτού. Yeah, colleagues, are you ready? So can we vote for... Ναι, αδελφοί, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Mm. Περνάμε τώρα στην πραγματική ψηφοφορία. Η γνωμοδότηση του Ρόπερτ Τζίλε, πλαίσιο ελέγχου των ξένων επενδύσεων, τροπολογία 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 97 και 177 υπέρ κατά να τις επαληθεύσουμε για αυτή την ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, ποια είναι η θέση του ΕΛΚ. Υπέρ. Όλοι υπέρ. Εγκρίνεται. 99 είναι συμβατή. Υπέρ, κατά, να την επαληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 100. Υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρες. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ή e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται ψηφοφορία 132 131 131 πέρας εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 138 υπέρ κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 150 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται, 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε, εντάξει. Δεν βλέπω χέρια. Πέρασε. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεργαστική Α υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω. Άρχεται η ψηφοφορία όμως. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 και λοιπές unblock υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 173 και 79 υπέρ. Κατά. Να τις επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στους ψηφορίες. Και εγκρίνεται. Και πάμε στο 176. 176 υπέρ, κατά, αποχές. Α, απορρίπτεται. 179 και άλλες δύο τροπολογίες και όλες μαζί υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Όχι, όχι, όχι, όχι μισό λεπτό. Καταπίπτει. Έχετε δίκιο. 178 υπέρ, κατά, αποχές. Είναι υπέρ το ΕΛΚ, ναι, ναι, ναι. Εγκρίνεται 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά Νομίζω ότι απολύτω αλλά θα κάνουμε έλεγχο για το 38. ο ψηφορίας. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 39. Είναι υπέρ. Το ΕΛΚ ναι. Άρα εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 44 ε, υπερκαταποχές εγκρίνεται, 45 υπερκαταποχές α, απορρίπτεται, το 2 υπερκαταποχές απορρίπτεται, 46 υπερκαταποχές εγκρίνεται, 47 υπερκαταποχές απορρίπτεται, Έλεγχο. Ψηφίζουμε για το 47. Πέρασε. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 4 48 υπερκαταποχές. κατά 49 υπερκαταποχές. Εγκρίνεται 50 υπερκαταποχές. Εγκρίνεται 51 υπερκαταποχές. κατά 52 υπερκαταποχές. Εγκρίνεται 5 υπερκαταποχές. Εγκρίνεται 53 υπερκαταποχές. κατά Συγγνώμη, καταπίπτει. 54 υπέρ εγκρίνεται. 55 υπέρ εγκρίνεται. 56 υπέρ εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά απορρίπτονται. 58 υπέρ εγκρίνεται. 59 υπέρ εγκρίνεται. 60 υπέρ εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά 6. Υπέρ, κατά, έλεγχος για το 6 ψηφίζουμε. Πέρασε. Και εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, η επόμενη έλεγχος για το 66 πέρας φιγορίας εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 όχι όχι δεν εγκρίνεται. Ναι, αλλά η Β Η Β συμβαστική. Αν είναι γιατί δύο λέει προς 69. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70. Υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 71. Συμβατή. Υπέρ κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Έλεγχος για το 71. Απορρίπτεται. Πέρασε. Απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά έλεγχος ψηφίζουμε Πέρασε. και εγκρίνεται 75 Εγκρίνεται. 77. Εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε ο βορείος. Εγκρίνεται ψηφίσουμε το κείμενο όπω τροποποιήθηκε. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίες. 38-8. Με τέσσερις αποχές συγχαρητήρια εισηγητά. Η επόμενη μας συνάντηση τώρα θα είναι στις 9 Τετάρτου, στις 3 η ώρα. Καλό Πάσχα. Πέρασε συνεδριάσεις. Και σας ευχαριστώ.